Ε, άρχεται η συνεδρίαση. Όπως ξέρετε, το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα είναι η ψηφοφορία για την αίτηση κατεπήγοντος πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου τροποποίηση του κανονισμού 1234 2007 ενιαίος κανονισμός ο ΚΟΑ με ε, τη θέσπιση ε, ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα. Ξαναδιαβάζω. Ε, πρόκειται για την θέση κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών. Η κυρία έχει, ο κύριος Ντεκάστρο έχει το λόγο. έχουμε ε, έχουμε ε, την ε, Επιτροπή Γεωργίας και μία τόπο θέτηση της Επιτροπής Αλίας. Ο κύριος Δεκάστρο έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, αγαπητοί φίλοι, Ξεκινάμε και πάλι ε, με τη συζήτηση του γαλακτοκομικού τομέα, ένα τομέα ο οποίος μας ανησυχεί πολύ και όπου η ε, γεωργοί ε, και οι αγρότες ε, ανησυχούν και εκδηλώνουν την ανησυχία τους. Έχουμε λοιπόν την υιοθέτηση της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ε, το γάλα ε, είτε υγρό είτε σε σκόνη και έχουμε διατάξεις και για τα τυριά αλλά θεωρούμε ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν και πρέπει να εξετάσουμε εάν θα πρέπει το άρθρο 186 της, ε, του, ε, του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ πρέπει να επεκταθεί και στο γάλα, δηλαδή να υπάρξει μία ε, διάταξη και ρύθμιση κατεπήγοντος χωρίς να περάσει από την κοινοβουλευτική εξέταση. Παρουσιάστηκε μία πρόταση της Επιτρόπου Fisher και θα ήθελα να ευχαριστήσω την επίτροπο που ήρθε στο Κοινοβούλιο μετά από το Συμβούλιο Γεωργίας που έλαβε χώρα στο Λουξεμβούργο για να μας αποδείξει το σεβασμό προς το σώμα μας και το εκτιμούμε. Εχθές ορισμένοι συνάδελφοι είχαν διατυπώσει κριτικές ε, λόγω της σοβαρής κατάστασης και είχαμε πει ότι το άρθρο 186 εμπόδιζε το Κοινοβούλιο να εκφραστεί πλήρως και ε, δίναμε ε, μία ευχέρεια ρυθμίσεως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ανησυχίες οι οποίες μας απασχολούν και πρέπει να σας πω κύριε Πρόεδρε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή έκανε σοβαρές προόδους και έλαβε υπόψη της ε, την γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου μας ε, εξήγησε πώς πρόκειται να χρησιμοποιήσει ε, το Ταμείο των 280 εκατομμυρίων ευρώ μας ανέφερε ότι υπάρχουν και διάφορα άλλα μέτρα τα οποία θα ληφθούν για την ιδιωτική αποταμίευση του τυριού και το το ποσό θα αυξηθεί στο επίπεδο που είχαμε ζητήσει ή στο ψήφισμα του Σεπτεμβρίου. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει σήμερα πιστεύω να υπερψηφίσουμε την αίτηση κατεπήγοντος γιατί οι κτηνοτρόφοι απαιτούν από εμά άμεση αντίδραση. Χάσαμε πολύ χρόνο, πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να επιταχύνουμε τη διαδικασία με, με Πρέπει λοιπόν εφόσον θα έχουμε συναπόφαση στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας να αναλάβουμε τα αναγκαία μέτρα. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για μία ψηφοφορία επί της αίτησης κατεπήγοντος, οπότε ο χρόνος παρεμβάσεως περιορίζεται σε τρία λεπτά. Κάποιος άλλος ζητά το λόγο, κάποιος είναι υπέρ ή κατά. Σας καλώ να εκφραστείτε. Yes, please. Ε, pan jest, pan jest za czy przeciw? Are you supporting? Είσαστε υπέρ ή κατά. Υπέρ ή κατά. Εγώ είμαι κατά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εδώ αναφερόμαστε στα θέματα του κατεπτύγοντος. Όχι ότι δεν χρειάζονται κατεπτύγοντα μέτρα, αλλά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει τα σωστά μέτρα και δεν θέλει ούτε είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την τωρινή κρίση του γάλακτος. Η Επιτροπή δεν επιλύει το πρόβλημα, αυτή είναι το πρόβλημα. Και γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε ότι ένα μέλος του προβλήματος το δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι επί μήνες δεν αντέδρασε κατά την κρίση. Το Φεβρουάριο η Επίτροπος μας είχε πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και η αγορά θα βελτιωθεί. Ας έχουμε υπομονή. Και ε, γι' αυτό ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι περιμένουμε την Επιτροπή να μας βοηθήσει. Δεν είναι σωστή οδός διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χθε δεν μπόρεσε να μας πει ε, γιατί θα πρέπει να διατεθούν δουν οι επιπρόσθετοι ε, πόροι. Μιλάμε ε, για αναδιάρθρωση ενώ μειώνονται συνεχώς οι γαλακτοκόμοι. Ε, πρέπει να ενισχύσουμε τους κτηνοτρόφους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αυξήσει τις επιδοτήσεις των εξαγωγών. Επίσης και για τα σούπερ μάρκετ δεν παρουσίασε μία λύση εχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οπότε δεν νομίζουμε ότι είναι σε θέση να λύσει σοβαρά την κρίση. Της δίνουμε μία επιταγή ελευτό χωρίς να ξέρουμε τι και πώς πρόκειται να πράξει. Ε, υπάρχει ένας βασικός λόγος επίσης ε, ότι ζητάμε από το Κοινοβούλιο να έχουμε περισσότερα δικαιώματα στον τομέα της γεωργίας και εδώ το πρώτο που κάνουμε πριν να έχουμε τα δικαιώματα αυτά είναι ε, να ε, μην ε, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει την κατάσταση στα χέρια του να την καθοδηγήσει και εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας σαν κοινοβουλευτικοί πρέπει να απαντήσουμε στην πρόκληση και να βοηθήσουμε τους γαλακτοπαραγωγούς με συνέπεια και συνέχεια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο κύριος Ντέσα 261 ζήτησε το λόγο. Κύριε Ντέσα, είσαστε υπέρ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι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 Συμφωνώ σε πολλά οποία είπε ο συνάδελφος αλλά δεν πρέπει να δώσουμε το λανθασμένο μήνυμα ή στου γαλακτοπαραγωγού που ζητούν μέτρα και γι' αυτό είμαι υπέρ τη διαδικασίας κατά τη διαδικασία αυτή πρόκειται να έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τα μέτρα και όπως είπε ο συνάδελφος υπάρχει η δυνατότητα με μία τροπολογία να περιορίσουμε τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δώσουμε δηλαδή εξουσιοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο για δύο χρόνια και να παραμείνει το κατεπήγον μόνο για μια συγκεκριμένη περίοδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, μόνο ένα άτομο κατεψήφισε, οι άλλοι υπερψήφισαν και όπως σας είπα ο λόγος περιορίστηκε εις ε, τα τρία λεπτά και τώρα ε, θέτω προς ψηφοφορία. Δεν πρόκειται να, υπάρχουμε, να έχουμε ονομαστική ψηφοφορία, άρα υπάρχει μία απλή ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ αυτής της αιτήσεως κατεπήγοντος. Ευχαριστώ. Ποιος είναι κατά. Ευχαριστώ. Ε, αποχές. Ευχαριστώ. αποφασίσει το κατεπήγον, δηλαδή υιοθετήθηκε η αίτηση κατεπήγοντος και σας υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία θα γίνει την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόταση η οποία έγινε προηγουμένως και οι τροπολογίες μπορούν να κατατεθούν μέχρι αύριο Τετάρτη. Σας παρακαλώ λοιπόν να σεβαστείτε ε, τον ε, χρόνο η συζήτηση θα γίνει απόψε. Σας υπενθυμίζω ότι η συζήτηση θα γίνει απόψε και οι ε, τροπολογίες μέχρι αύριο στις 10 πρέπει να έχουν κατατεθεί. Τώρα λοιπόν έχουμε τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την κλιματική αλλαγή και αναπτυσσόμενες χώρες στα πλαίσια της ε, διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών στην Κοπενχάγη σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Θέλω να παρακαλέσω τον Υπουργό του Περιβάλλοντος